Dear colleagues, συνάδελφοι, ας ξεκινήσουμε την συνεδρίασή μας πρώτα απ' όλα με την έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Αυτή δεν συμπεριλαμβάνει τον δημοσιονομικό διάλογο με τον ε, Υπουργό Οικονομικών της Λετωνίας και προεδρεύοντα του Συμβουλίου ΕΚΟΦΗΝ διότι λόγω της συνάντησης του Eurogroup για, τις, για την παράταση του προγράμματος της Ελλάδας και τις συνεχιζόμενες διπλωματεύσεις δεν θα μπορέσει να είναι σήμερα στην Επιτροπή μας ο Υπουργός Αναβάλλεται λοιπόν αυτή η συνάντηση και ο οικονομικός διάλογος. Άλλες ανακοινώσεις. Πρώτα απ' όλα μία θετική. Επετεύχθη πολιτική συμφωνία στον τριμερή διάλογο για τον κανονισμό, για την υποβολή εκθέσεων και τη διαφάνεια στις ε, οικονομικές συναλλαγές. Πολύ καλό αποτέλεσμα. Έχουμε την πρώτη συμφωνία για τον παρατραπεζικό τομέα από τους συνομοθέτες και το κείμενο της συμφωνίας περιλαμβάνει πολλά από τα σημεία που το Κοινοβούλιο ήθελε να συμπεριληφθούν στο τελικό νομοθετικό κείμενο. Σε χαρητήρια λοιπόν στον εισηγητή, τη διαπραγματευτική ομάδα και τη γραμματεία. Επίσης επισήμως να ανακοινώσω ότι πετεύχθη συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του, Συμβουλίου του Κοινού Μηχανισμού Εξυγίανσης για τις διαδικασίες λογοδοσίας και δημοκρατικής επίβλεψης σε σχέση με τις αρμοδιότητες που ανατίθενται στο Συμβούλιο του Κοινού ε, μηχανισμό εξυγίανσης βάσει των κανόνων της. Ε, επετέχθη λοιπόν συμφωνία. Το κείμενο θα αποσταλεί και στη διάσκεψη των Προέδρων που είχε δώσει την αρχική εντολή για τις διαπραγματεύσεις. Δεύτερος γύρος του τριμερούς διαλόγου για τον κανονισμό συγκριτικής αξιολόγησης στις 22 Ιουνίου. Επετέχθη πρόοδο σε αυτή τη συνάντηση. Αλλά και πάλι χρειάζεται πολλή δουλειά Οπότε θα συνεχίσει επί Λουξεμβουργιανής Προεδρίας η σύγχρονη συζήτηση. Και επίσης βρισκόμαστε κοντά στην τελική συμφωνία για την ε, οικονομική διαμεσολάβηση και μάλλον ο τελικός γύρος θα λάβει χώρα την επόμενη Τρίτη. Σας ευχαριστώ. Α, ναι. Αντιπροσωπεία της Επιτροπής μας. Επισκέφτηκε τη Μαδρίτη την περασμένη εβδομάδα. Ήταν ιδιαίτερα επικοδομητική, εντατική και ενδιαφέρουσα η συνάντηση με τις Ισπανικές αρχές, με τις οποίες συζητήσαμε ένα ευρύ θεμάτων μεταξύ των οποίων όχι μόνο η ισπανική οικονομική και δημοσιονομική κατάσταση, αλλά και η συνεισφορά της Ισπανίας στη δουλειά των πέντε προεδριών. υπάρχει μεγάλο βαθμό σύγκληση με τα όσα επιθυμεί και το Κοινοβούλιο σε αυτή την περίπτωση. Σα ευχαριστώ και τώρα να καλωσορίσω την Ντανιέλ Νούι, πρόεδρο του Υποπτικού Συμβουλίου τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στα πλαίσια του κοινού εποπτικού μηχανισμού. Πρώτα δημοσια, πρώτη δημόσια ακρέωση για τη φετινή χρονιά, γιατί ο κοινωνικό εποπτικό μηχανισμό προβλέπεται στη Διεθνική Συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και Συμβουλίου και βάσει τη απόφαση των συντονιστών του Μαΐου η κυρία Νούι έχει προσκληθεί στη δημόσια κρόασή μας σήμερα, ιδίως για τα εξής ζητήματα. Το Anacredit, ένα σύστημα που ξεκίνησε από το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Κεντρικών Τραπεζών για τα οικονομικά στοιχεία των τραπεζικών ε, ιδρυμάτων εκτός τραπεζικού τομέα, των κεφαλιακικών απαιτήσεων και μια σειρά από άλλα ζητήματα. Έχετε το λόγο, Ντανιέλ. Ευχαριστώ, καλημέρα σα. Ε, είναι χαρά που ξαναβρίσκομαι εδώ στην ΚΟΝ, στι αγωγικέ μου παρατηρήσεις. Θα σας κάνω μια συνόψη της κατάστασης στον τραπεζικό τομέα που επιτηρεί ο ενιαίο μηχανισμός επιτήρηση και θα μιλήσω για τα προγράμματα που μας απασχολούν τώρα. Θα συζητήσω επίση τα θέματα που μου ζητήσατε να συζητήσω, δηλαδή οι κεφαλικές απαιτήσει για τις τράπεζες, το ΣΡΕΠ και ε, το ANA Credit. Θα μιλήσω λιγάκι και για τη συνεργασία με τον ενιαίο μηχανισμό εξυγίανσης. Λοιπόν, να ξεκινήσω με μια επισκόπηση του τραπεζικού τομέα. Οι ευρωπαϊκές ε, τράπεζες, οι τράπεζες της Ευρωζώνης αντιμετωπίζουν τα θέματα του παρελθόντος από την οικονομική κρίση προσαρμοζόμενες επίσης και στο κανονιστικό και λειτουργικό περιβάλλον που αλλάζει. Η συνολική αποτίμηση έδειξε ότι χρειάζεται πολύ διαφάνεια και την επιφέραμε αυτή τη διαφάνεια και έδειξε ότι ο τραπεζικός τομέας είναι καλά εξοπλισμένος για να αντιμετωπίσει τις πιο πιθανές αρνητικές επιθέσεις κλειδονισμού. Ωστόσο, έχουμε ορισμένα προβλήματα. Οι τράπεζε τη Ευρωζώνη έχουν σχετικά αδύναμη κερδοφορία. Αυτό έχει να κάνει με το πόσο ευαίσθητη και άνηση είναι η ανάκαμψη και επίσης το ότι έχουμε ένα περιβάλλον ε, χαμηλών επιτοκίων που πιέζει τα κέρδη τους. Ε, ναι, μεν υπάρχουν ε, ορισμένα στοιχεία ότι βελτιώνει η κατάσταση, αλλά πρέπει ίσω να γίνουν περαιτέρω προσαρμογέ στον τρόπο λειτουργία του. Μία δεύτερη πρόκληση είναι ότι έχουν πολλά προβληματικά στοιχεία ενεργητικού ορισμένε τράπεζε που δεν του επιτρέπει να δανείζουν αρκετά. Είναι λοιπόν ιδιαίτερα πιεστικό αυτό για τι τράπεζε που λειτουργούν σε ένα πιο ευάλωτο οικονομικό περιβάλλον στι χώρε του. Το πρόβλημα των μη εξυπηρετουμένων δανείων Χρειάζεται μια σφαιρική προσέγγιση, αλλά δεν υπάρχει μια λύση για όλου, διότι τα προβλήματα αυτά έχουν να κάνουν με διαφορετικέ αιτίε ε, συμπεριλαμβανομένων και των γενικών οικονομικών συνθηκών, κακών τραπεζικών πρακτικών, αδύναμου νομικού πλαισίου για την ανάκτηση των χρεών και έλλειψη δυνατοτήτων του δικαστικού συστήματος. Μερικά από αυτά τα αίτια ξεπερνούν την εντολή του SSM. Συνολικά η ε, χαμηλή κερδοφορία και τα πολλά προβλήματα του παρελθόντος με ορισμένα στοιχεία του ενεργητικού εξακολουθούν να επηρεάζουν τις τράπεζες για να δημιουργήσουν και το κεφαλικό απόθεμα, κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας και να δώσουν πιστό στην πραγματική οικονομία. Τώρα να δούμε ποια είναι τα βασικά μας προγράμματα και αποφάσεις από τότε που σας είδα τον Μάρτιο. Το Μάρτιο ανέφερα ότι η διαδικασία δημιουργίας του SSM είχε πλήρως και επιτυχώς ολοκληρωθεί. Παρ' όλα αυτά χρειαζόμαστε να δουλέψουμε ακόμη για να φτάσουμε σε μια ε, σταθερή κατάσταση και μαθαίνουμε κάθε μέρα. Ορισμένα θέματα θα πάρουν τον χρόνο τους, όπως για παράδειγμα μια κοινή εποπτική κουλτούρα εντός του SSM. Αυτό είναι καθημερινή προσπάθεια και είμαι πεπισμένη ότι σύν χρόνο θα δώσει τα ε, επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Με βάση αυτό το πλαίσιο έχουμε αναλάβει την εξάμηνη ε, αναθεώρηση των προτεραιοτήτων μας για να είναι πάντα ενημερωμένες, για να λάβουμε υπόψη τις πρόσφατες εξελίξεις και την ε, αποτίμηση που κάνουμε των βασικών κινδύνων. Αυτές οι εξελίξεις ε, αναλαμβάνουν τις, περιλαμβάνουν τις αναγκαίες προσαρμογές για να επιτύχουμε το BRRD, MREL και TLAC την ε, ποιότητα του κεφαλαίου των τραπεζών ιδιότερα σε σχέση με τα αναβαλώμενα ε, στοιχεία φορολογίας και τις ε, φορολογικές πιστώσεις και εκτόσεις και την αβεβαιότητα όσον αφορά την παρατηνόμενη κατάσταση χαμηλών επιτοκίων. Προσαρμόσαμε ελαφρώς τις προτεραιότητές μας και αυτό θα αντανακλαστεί στις ενέργειές μας. Να στραφώ τώρα στα δύο πρώτα θέματα που προτείνατε ε, πρώτα απ' όλα την, ε, τις κεφαλαϊκές απαιτήσει και το ΣΡΕΠ. Στόχος μας μέσω αυτών των κεφαλαϊκών ε, απαιτήσεων είναι να δούμε ποιες τράπεζες είχαν έλλειψη. Για να υπενθυμίσω, η σφαιρική αποτίμηση βρήκε σε 24 τράπεζες έλλειψη κεφαλαίου, συνολικά 24,6 δις. Κατά τη διάρκεια του 2014 οι τράπεζες μπόρεσαν να βρουν 18,6 δισεκατομμύρια νέου κεφαλαίου. Κατά συνέπεια, μερικές τράπεζες έχουν ήδη επιλύσει το πρόβλημα ελλείψεων κεφαλαίου πριν τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της σφαιρικής αποτίμησης τον περασμένο Οκτώβριο. Περαιτέρω, οι τράπεζες ε, χρειαζόταν να καλύψουν τις ελλείψεις κεφαλαίου εντός 6 μηνών ή 9 μηνών μετά την ε, δημοσίευση των αποτελεσμάτων εφόσον ήταν από τα stress test, τα test αντοχής αυτές οι ε, διαπιστωθήσεις ε, ε, ελλείψεις. Οπότε τον Αύγουστο είναι η προθεσμία. Αρχές Ιουνίου περισσότερες τράπεζες είχαν καλύψει αυτές τις ελλείψεις. Και από τις λίγες που έχουν ακόμη προβλήματα, οι περισσότερες θα μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες τους πριν τη λήξη της προθεσμίας. Τώρα, για να δούμε τώρα το ΣΡΕΠ, e που όπως ξέρετε καθορίζει για κάθε τράπεζα τις συγκεκριμένες κεφαλαϊκές απαιτήσει για τη συγκεκριμένη τράπεζα στα πλαίσια του πυλώνα 2. Η έγκριση των αποφάσεων του ΣΡΕΠ για το 2015 για όλες τις τράπεζες έχει ολοκληρωθεί. Αυτές οι αποφάσεις λήφθηκαν στις αρχές του 2015 στη βάση των εθνικών προσεγγίσεων ΣΡΕΠ διότι αυτή η εργασία έγινε το 2014 και συμπληρώθηκε από τα αποτελέσματα της σφαιρικής αποτίμησης του SSM δεν ήταν μόνο θέματα έλλειψη κεφαλαίων, γιατί πρέπει να δούμε και πώς θα καλύψουμε ακόμη και για καλά κεφαλαιοποιημένες τράπεζες τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Από φέτος θα παρακολουθήσουμε, θα ακολουθήσουμε μάλλον για πρώτη φορά μια ενιαία προσέγγιση ΡΕΠ. Αυτό είναι βασικό στοιχείο για τον ενιαίο επιτηρητή και έχει στόχο να υπάρχει συνεπής αντιμετώπιση των σημαντικών πιστοτικών ιδρυμάτων σε όλους τους τομείς που καλύπτει το SSM. Για να υπάρχει μια συνεπής εφαρμογή της μεθοδολογίας REP, κάνουμε μια σε βάθος οριζόντια ανάλυση και οι αποτιμήσεις REP θα προσαρμοστούν με βάση το αποτέλεσμα αυτής της οριζόντιας ανάλυσης. Πρέπει όλοι να αναγνωρίσουμε, ωστόσο, ότι η συνέπεια στις εποπτικές προσεγγίσεις θα είναι πιο αποτελεσματική αν όλοι οι θεσμοί που υπόκεινται στο SSM έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις όσον αφορά το ρυθμιστικό πλαίσιο από την κατάσταση αυτή. Ακόμη απέχουμε από ικανοποιητική κατάσταση γιατί υπάρχουν διαφορετικές, σημαντικές διαφορές στους εθνικούς κανονισμούς για τις τράπεζες εντός του SSM και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα μόνο στα λόγια έχουμε ένα ενιαίο σύνολο κανόνων για τις τράπεζες, όχι στην πράξη. Οπότε για να δούμε ποια είναι η κανονιστική αντιμετώπιση των κεφαλαίων. Αυτό μας φέρνει στις λεγόμενες εναλλακτικέ λύσεις ή τα εθνικά μέτρα. Ένα από τους βασικούς στόχους του Βασιλεία 3 ήταν να έχουμε ένα πιο ανθεκτικό τραπεζικό τομέα, αυξάνοντας και την ποιότητα και την ποσότητα του κεφαλαίου. Όπως ξέρετε, η Βασιλεία 3 εγκρίθηκε στην Ευρώπη μέσω του πακέτου CRDIV-CRR. Και το Βασιλεία 3 και το πακέτο CRDIV-CRR περιλαμβάνουν μεταβατικές διατάξεις, ούτως ώστε να μπορέσει ο τραπεζικός τομέας να ανταποκριθεί στις υψηλότερες κεφαλαϊκές απαιτήσει μέσω ε, διατήρησης κάποιων κερδών και αύξηση κεφαλαίου, αλλά συνεχίζοντας να δίνει ε, στην οικονομία. Το πακέτο αυτό επέτρεψε στις αρμόδιες αρχές να αποφασίσουν πώς θα εφαρμόσουν αυτές τις ε, μεταβατικές διατάξεις, αλλά αυτό είχε ως αποτέλεσμα άνηση εφαρμογή τους μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών. Από τότε που το ECB έχει γίνει η αρμόδια αρχή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δηλαδή, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να λαμβάνει εποπτικές αποφάσεις προς το ε, βέλτιστο συμφέρον της Τραπεζικής Ένωσης. Με αυτήν την προσπάθεια, λοιπόν με αυτό το εγχείρημα στο μυαλό, ξεκινήσαμε μια προσπάθεια να εναρμονίσουμε όπου θα πρέπει και με πολύ αυστηρό τρόπο να υπάρχει λοιπόν εναρμόνιση και των μεταβατικών και των μονίμων εναλλακτικών λύσεων και επιλογών που έχουν οι κυβερνήσεις. Αυτές οι επιλογές και οι εθνικές αποφάσεις συζητιούνται τώρα σε συντονισμό με τις εθνικές αρμόδιες αρχές και την ε, Τραπεζική Ένωση για να προωθήσουμε την ολοκλήρωση και την δημοσιονομική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Να συζητήσω ένα άλλο θέμα που μου θέσατε, το Anacredit, την πρωτοβουλία Anacredit. Αυτή η προσπάθεια, αυτό το εγχείρημα ξεκίνησε πριν ξεκινήσει το SSM. Αρχικός στόχος ήταν να δημιουργηθεί ένα βασικό κανόνων εναρμονισμένων λεπτομεριακών στοιχείων που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από διάφορε κεντρικέ τράπεζε για διάφορου σκόπου, όπω για παράδειγμα νομισματική πολιτική και λειτουργίε, διαχείριση κινδύνου, χρηματοπιστωτική σταθερότητα, έρευνα και στατιστικά. Καθ' όλη τη διάρκεια του σχεδιασμού και της ε, έναρξης αυτής της ε, ε, προσπάθεια, είχαμε υπόψη μα επίση την ανάγκη να μειωθούν οι ανάγκε υποβολή στοιχείων. Η πρώτη φάση αυτού του προγράμματος Anacredit προβλέπεται να λειτουργήσει μέχρι τις αρχές του 2018. Τώρα στοχεύουμε στις, στα δάνεια που δίνουν σε επιχειρήσεις και τράπεζες με κατόφλι 25.000 ευρώ. Θα μας επιτρέψει λοιπόν να αναλύσουμε πώς δανείζουμε στις μικρομέσες αργότερα, που προβλέπουμε να είναι το 2020, θα δούμε και τα ενυπόθηκα δάνεια των οικοκυριών, και τα δάνεια προς τους λεγόμενους ε, μεμονωμένους ε, ιδιοκτήτες, δηλαδή αυτούς που είναι οι μόνοι ιδιοκτήτες μιας επιχείρησης ή αυτοπασχολούμενοι. Αυτό θα γίνει όμως μόνο σε ανωνυμοποιημένη βάση και θέλω να υπογραμμίσω ότι δεν θα συλλεγούν ευαίσθητα στοιχεία όπως οικογενική κατάσταση ή θρησκεία ή οποιαδήποτε άλλη ευαίσθητη πληροφορία. Δεν θα συλλεγούν τέτοια ευαίσθητα στοιχεία παρόλα αυτά παρά το ότι ξεκινήσαμε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πριν έχει εποπτικά καθήκοντα η Κεντρική Τράπεζα, οι νέες ε, λειτουργίες εποπτείας θα ωφεληθούν. Το ανακρέδιτ μας δίνει συγκρίσιμα στοιχεία σε υψηλό επίπεδο λεπτομέρειες, ιδιαίτερα όσον αφορά την κατανομή του χαρτοφυλακίου των τραπεζών ανά ε, δηλαδή ποια είναι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια κτλ και οι δείκτες και οι αναλύσεις που θα προωθήσουν τους επιτηρητές για παράδειγμα για να έχουμε σταθμισμένη εκτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και για να βοηθήσουμε τις τράπεζες στην εποπτική λειτουργία. Για να καταλήξω τώρα να σας πω ποια είναι η αλληλεπίδραση μεταξύ όλων των εποπτικών αρχών και των αρχών εξυγίανσης. Είμαι πεπισμένη ότι το SSM θα κερδίσει πολλά έχοντας ε, μια ισχυρή SRM στο πλευρό της. Γι' αυτό δεσμεύομαι να δημιουργήσω μια πολύ στενή συνεργασία μεταξύ του SSM και του SRM. Αυτό θα είναι αμοιβαία εποφελές Θα μας βοηθήσει να μειώσουμε τη γραφειοκρατία για το τραπεζικό σύστημα και να μην λαμβάνουν ε, αντιφατικά μηνύματα οι τράπεζες. Η συνεργασία μεταξύ SSM και SRM θα περιγραφεί σε ένα μνημόνιο συνεννόησης το οποίο θα περιγράφει τις ροές πληροφοριών μεταξύ των δύο αρχών. Ήδη σε αυτή τη φάση η Κεντρική Τράπεζα και το SRB ανταλλάσσουν πληροφορίες όπως προβλέπεται στο νομικό πλαίσιο. Η συνεργασία με βάση αυτό το μνημόνιο έχει ξεκινήσει. Το μνημόνιο που είναι σε φάση διαμόρφωσης και συνεργαζόμεθα για διάφορα θέματα ιδιαίτερα όσον αφορά τη μηχανοργάνωση. καταλήγοντα. Πολλά έχουν ήδη επιτευχθεί από τότε που ξεκίνησε το SSM, αλλά έχουμε μπροστά μας ε, διάφορες ακόμη προκλήσεις. Η ευθυγράμμιση των εποπτικών προσεγγίσεων και πρακτικών σε όλο το μήκος του SSM για να έχουμε υψηλού επίπεδου και αυστηρά ε, στάνταρ είναι μία από τις προτεραιότητές μας. Προς αυτή την κατεύθυνση φέτος ξεκινήσαμε μία σφαιρική αναθεώρηση των εσωτερικών προτύπων για κεφαλαικές απαιτήσεις των τραπεζών και για την ε, εκ των προτέρων ε, εποπτεία και στοχεύουμε να έχουμε συνεπή αποτελέσματα της ε, εποπτικής μας δραστηριότητας και έντασης και να δημιουργήσουμε έντονη συνεργασία εντός και εκτός του SSM. Τέλος, προσβλέπουμε στην κατάληξη της νομοθετικής διαδικασίας για την διαθροτική μεταρρύθμιση των τραπεζών Πέρα από το περιεχόμενο αυτής της κατάληξης, η ίδια κατάληξη θα άρει την ισχύουσα τώρα αβεβαιότητα και θα επιτρέψει στις τράπεζες να εξελίξουν, να εφαρμόσουν το μακροπρόθεσμο τρόπο λειτουργία του. Και ελπίζουμε ότι το Κοινοβούλιο θα παίξει το ρόλο του, τόσο ώστε αυτό το νομικό πλαίσιο να επιτρέπει μια, ομόφορμη, μια ομοιόμορφη εφαρμογή του κανονισμού εντό του SSM. Σε ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σα. Ευχαριστούμε πολύ. Είμαι βέβαιος ότι το Κοινοβούλιο θα κάνει ό,τι μπορεί για να επιτρέψει να ζητήσει ομοιόμορφη εφαρμογή. Και τώρα η ομιλητέ. Γεώργιος Κύρτσος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι για το τι συμβαίνει στον τραπεζικό τομέα στην Ισπανία και Πορτογαλία μετά από επίσκεψη στη Μαδρίτη νομίζω ότι διαπιστώθηκε πολύ καλή λειτουργία των Ισπανικών τραπεζών, έλυσαν πολλά τους προβλήματα που είχαν στο παρελθόν. Απ' την άλλη, μπορεί να υπόκεινται σε επιπτώσεις από την ελληνική κρίση, γιατί ξέρετε ότι υπάρχει και τραπεζική και οικονομική κρίση στην Ελλάδα πράγμα το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε κρίση εμπιστοσύνη στο Ευρωζώνη ή σε τμήματά της. Θα μπορούσατε μήπως να μας συνοψίσετε ως πρόεδρος του ενιαίου Ποπτικού μηχανισμού ποια είναι τα ισχυρά σημεία του ισπανικού και πορτογαλικού τραπεζικού τομέα και τι πρέπει να ενδυναμώσουν και να προσέξουν. Ευχαριστώ. Ναι. Ευχαριστώ για το ερωτήσει σας. Οι χώρες που αναφέρατε, όπως και άλλες, όταν γίνεται πραγματική αναδιάρθρωση τραπεζών, έχουν καλά αποτελέσματα Δεν υπάρχει λοιπόν κανένας λόγος να πιστέψουμε ότι επειδή αποπτεύονται από το SSM τώρα, το ΚΕΜ e θα υποφέρουν από επιπτώσεις από την ελληνική κρίση. Δεν αναμένουμε τέτοιες επιπτώσεις για τις ευρωπαϊκές τράπεζες ή τις τράπεζες υπό το ΚΕΜ. Ελίζα Φερέιρα. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε σήμερα και για όλες τις πληροφορίες που μας δίνετε. Αναφέρατε τη σχέση μεταξύ αποπτίας και εξυγένσης. Ωστόσο, ενημερωθήκαμε από την κυρία Κέρνινγκ ότι υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση στην ε, μεταφορά της οδηγίας για τις κεφαλικές απαιτήσεις. Πόσο αποτελεσματική λοιπόν είναι η διαδικασία της εποπτείας όταν ζητάτε περισσότερα κεφάλαια ή τη αφήνεια για τους όρους που διέπουν τις αυξήσεις των κεφαλαίων σε σχέση με τον πληθωρισμό και την κάλυψη των κινδύνων. Ποια είναι η φιλοσοφία σας, η συλλογιστική σας όταν χρησιμοποιείτε αυτά τα χρονοδιαγράμματα τις εθνικές επιλογές, όλες αυτές τις δυνατότητες μετάβασης. Ποια είναι η φιλοσοφία σας, ποιες οι μεριμνές σας και πώς ερμηνεύετε τις ενδεχόμενες καθυστερήσεις και για, το, ε, για, τους, ε, για την ισοτιμία των κανόνων ως προς την κοινή εποπτεία. Αυτή είναι η ερώτησή μου προς τη μήνυ. Κοιτάξτε, συμφωνώ με την άποψή σας ότι η οδηγία για την εξυγίανση και τη διάσωση πρέπει να μεταφερθεί στο δυνατόν συντομότερα. Ή δυνατόν έπρεπε να είχε μεταφερθεί στις αρχές αυτής της χρονιάς. Οι επιπτώσεις για τους επόπτες είναι ότι αντί να έχουμε κοινά εργαλεία ή μια κοινή γλώσσα όπως προβλέπει η οδηγία, Αναγκαζόμαστε να μελετούμε όλα τα εθνικά συστήματα των χωρών που δεν έχουμε μεταφέρει πλήρω στην οδηγία. Δηλαδή, χρειάζονται περισσότερε γνώσει, περισσότερο χρόνο που θα μπορούσαν να έχουν δαπανηθεί καλύτερα σε υποπτικέ διαδικασίε. Δεν γίνεται αδύνατη λοιπόν η προσπάθειά μα, γίνεται όμω πολύ πιο περίπλοκη. Αυτό ισχύει για τις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει εναρμόνιση. Διότι η οδηγία έχει μεταφερθεί πολύ καιρό πριν τον ενιαίο αποπτικό μηχανισμό. Υπάρχουν διαφορετικές διαδικασίες μεταφοράς σε κάθε νομοθεσία, σε κάθε κράτος ή μπορεί να υπάρχει πολύ περιθώριο ελαστικότητας λόγω της χρήσης των εθνικών επιλογών. Πρέπει να έχουμε εναρμονισμένους κανόνες για να υπάρχει εναρμονισμένη εποπτεία. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ναι, αλλά η μη μεταφορά μπορεί να φέρει τελικά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για κάποιες τράπεζες. Αυτό είναι το πιο ανασχετικό. Δεν είμαι βέβαια. Δεν είμαι βέβαια ότι προσφέρει πλεονεκτήματα η καθυστέρηση. Απλώς γίνεται πολύ πιο δύσκολη η δική μας δουλειά. Αυτό είναι το προφανές. Και όπως είπατε πρόεδρε, θα είναι ακόμη πιο σημαντικό το 2016. Αυτό που συμβαίνει όμως, ήδη μέρος της οδηγίας ε, έχει υλοποιηθεί από φέτος και όταν η οδηγία δεν υλοποιείται πρέπει να χρησιμοποιούμε τους εθνικούς νόμους. Κάποιες φορές βρίσκονται πολύ κοντά στην οδηγία, κάποιες φορές δεν υπάρχουν ή υπάρχουν και είναι τόσο διαφορετική από αυτά που προβλέπει η οδηγία που τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο δύσκολα. Πρόεδρος. Ευχαριστούμε και πρέπει να παροτρύνουμε ε, τα κράτη-μέλη να κάνουν τη μεταφορά στο δυνατόν πιο γρήγορα. Με συγχωρείτε. Με Επόμενος ο μιλητής, ο κύριος Όλο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Μετά τον εποπτή την θέση ενισχύ του εποπτικού μηχανισμού. Τώρα εποπτεύονται κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών, όχι μόνο εθνικών ιδρυμάτων, αλλά φαντάζομαι και οι δοσοληψίες που κάνουν τραπεζικοί όμιλοι. Και εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι η εποπτεία των δοσοληψιών. Έχω μία θεωρητική ερώτηση. Αλλά υπάρχει και ένα πρακτικό παράδειγμα. Αν σε μία χώρα που καλύπτει ο εποπτικός μηχανισμός, εάν μία τράπεζα πουληθεί και αρχίσει συζήτηση για τον, την ακριβή της τιμή πώλησης και υπάρξουν αμφιβολίες ως προς το κατά πόσον έγινε καλή την πίστη η πώληση, σε ποιο βαθμό τότε μπορούμε να αναμένουμε παρέμβαση από την έκτη και τον εποπτικό μηχανισμό. Αυτό ήταν το πρώτο ερώτημα. Το δεύτερο. Πώς κατανέμονται οι αρμοδιότητες μεταξύ έκτα από τη μία και εθνικών εποπτικών μηχανισμών από την άλλη. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε λιγάκι. Ευχαριστώ. Για τις πωλήσει τραπεζών από ό,τι κατάλαβα ενδιαφέρεστε για την τιμή. Εμείς οι επόπτες δεν ασχολούμαστε με την τιμή. Είμαστε υπεύθυνοι μόνον για το λεγόμενο qualifying holding, δηλαδή αγοραστές των τραπεζών, αν είναι διατεθειμένοι και ικανοί να λειτουργήσουν σωστά την τράπεζα, τότε δεχόμαστε αυτούς τους μετόχους ως νόμιμους. Αλλά το αποτέλεσμα της απόρρι... μιας απόρριψης θα ήταν ότι μπορεί να αποφασίσουμε ότι οι νέοι αυτοί equity holders δεν θα έχουν δικαιώματα ψήφου. οι μέτοχοι. Εάν δεν θεωρηθούν κατάλληλοι για αυτή την τράπεζα. Αυτό είναι ο μόνος ρόλος που παίζουμε. Όπως και πριν εξάλλου με τους εθνικούς επόπτες. Τώρα είναι το ΚΕΜ Επιταρωτήσατε πώς χωρίζονται, πώς κατανέμονται οι δικαιοδοσίες, οι αρμοδιότητες μεταξύ ΕΚΤ και εθνικών εποπτών. Μερικές δικαιοδοσίες και αρμοδιότητες σαφώς είναι στα χέρια του ΚΕΜ, δηλαδή και των εθνικών εποπτών και της ΕΚΤ αν χρειαστεί ανακεφαλαιοποίηση ας πούμε. Άλλες, σαφώς επίσης, είναι ακόμη στα χέρια των εθνικών εποπτών όπως το ξέπλυμα βρωμίκου χρήματος ας πούμε. Και υπάρχει επίσης και μία γκρίζα ζώνη για την οποία πρέπει να πάρουμε νομικές συμβουλές αναπερίπτωση από τους δικηγόρους μας της ΕΚΤΑ ας πούμε εθνικές επιλογές αν έχουν μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο και άρα είναι στα χέρια των εθνικών αρχών. Από τον Νοέμβριο όμως αυτά τα αναλαμβάνει το ΚΕΜ αλλά αν έχουν μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο πριν από τον καθορισμό του ΚΕΜ μπορούμε να θεωρήσουμε ότι παρόλα αυτά είναι στα χέρια του, του ΚΕΜ ή όχι. Αν επρόκειτο για εθνικές επιλογές, τότε θα ίσχυε αυτό. Ο κανονισμός έρχεται πρώτος. Εφαρμόζεται κατευθείαν η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αν είναι μεταφορά οδηγίας δεν είναι σαφές. Αυτό είναι μία από τις δυσκολίες της λειτουργίας του ΚΕΜ για τον πρώτο χρόνο. Πρέπει να είμαστε νομικά σίγουροι όταν παίρνουμε αποφάσεις. Α, σιγά σιγά μαθαίνουμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Επόμενος μιλητής, ο κύριος Ούρμπαν από την ΚΟΕ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Προτείνετε και συμβουλεύετε τις ελληνικές τράπεζες να μειώσουν την έκθεσή τους στην, ε, στο, στα εθνικό, ελληνικό δημόσιο χρέος, στα ελληνικά ομόλογα. Αυτή είναι η ερώτησή σας. Τι έννοια έχει αυτό όταν το ελληνικό κράτος είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να στηρίξει τις ελληνικές τράπεζες σε περίπτωση πτώχευσης. Με αυτό το μορφό, εάν ε, πέσει το ελληνικό κράτος, πέφτει και ο ελληνικός ε, τραπεζικός τομέας. Άρα είναι λίγο περίεργο να απαιτείται από τον ελληνικό τραπέζι, τραπεζικό τομέα να δυσχεράνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση ρευστότητας της ελληνικής κυβέρνησης. Δεν έχει λοιπόν καμία έννοια αυτό εάν θέλουμε να αποφύγουμε την ε, πτώχευση των ελληνικών τραπεζών. Πώς το αντιμετωπίζετε αυτό. Καταρχάς να πω ότι έχουμε θαυμάσια συνεργασία με τους Έλληνες επόπτες που είναι μέλη του εποπτικού μας συμβουλίου, είναι πολύ καλοί, έχουν κάνει καταπληκτική δουλειά για να αναδιοργανώσουν, να αναδιαρθρώσουν τον ελληνικό τραπεζικό τομέα τα τελευταία χρόνια και όπως τα είδατε οι ελληνικές τράπεζες τα έχουν πάει αρκετά καλά <clears throat> κατά την ε, συνολική αποτίμηση. Έχω συζητήσει επανειλημμένα την κατάσταση του ελληνικού τραπεζικού τομέα και ενώπιον της ΕΚΟΝ. Δεν έχω τίποτα να προσθέσω. Και προσβλέπω, όπως και οι συνάδελφοί μου, προσβλέπω στην ε, παρατήρηση λευκού καπνού ότι θα υπάρξει δηλαδή συμφωνία σε πολιτικό επίπεδο. Μέχρι να γίνει αυτό Κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε ως επιτηρητές, παρατηρούμε την ε, ρευστότητα και την φερεγγιότητα. Αυτή είναι η συνήθις εργασία μας. Ο κύριος Γκίγκολτ. Α, όχι, εσείς παρακαλώ. Με συγχωρείτε, αλλά δεν νομίζω ότι μου απαντήσατε, λέει ο κύριος Σούρμπαν, στην πρώτη μου ερώτηση. Συμβουλεύετε τις ελληνικές τράπεζες να μειώσουν την έκθεσή, της, την έκθεσή τους στο δημόσιο ελληνικό χρέος. Αυτή ήταν η ερώτησή μου. Το συμβουλεύετε. η ε, κυρία Νούη, εμείς δεν δίνουμε συμβουλές ούτως ή άλλως. Δεν είναι η δουλειά μας. Εμείς εκτιμούμε καταστάσεις με βάση το νομικό πλαίσιο και άλλα στοιχεία και παίρνουμε αποφάσεις. Οι αποφάσεις μας δεν είναι δημόσιες. Δεν μπορώ να τις σχολιάσω. Δεν σχολιάζω τις αποφάσεις που μπορεί να έχουν ληφθεί όσον αφορά τις ελληνικές τράπεζες. Ευχαριστώ, Σβέν Γκίγκολτ. Καλώς ήρθατε και σας ευχαριστούμε πολύ για τη δουλειά σας, για την ε, ανοικοδόμηση όλου αυτού του συστήματος, όλου αυτού του μηχανισμού. Προχωρά ε, ο μηχανισμός και αυτό είναι θετικό για την Ευρώπη, είναι μια καλή είδηση. Έχω κάποιες ερωτήσεις κι εγώ όμως. Σε ό,τι αφορά τη μεθοδολογία της αξιολόγησης κινδύνου. Καταλαβαίνω ότι δεν κάνετε διάκριση μεταξύ μικρότερων ιδρυμάτων και μεγαλύτερων. Μπορείτε να ενημερώσετε το Κοινοβούλιο ή να το ενημερώνετε πιο συστηματικά για τη διάκριση που κάνατε μεταξύ μεγαλύτερων και μικρότερων ιδρυμάτων. Αυτό είναι μέρος του κανονισμού. Αλλά δεν νομίζω ότι η διάκριση που γίνεται τώρα συνάδει με την αρχή της αναλογικότητας. Επίσης, έτσι όπως το εξηγήσατε, το ανακρέντιτ και επειδή δημιουργήθηκε πριν από τη δημιουργία του ενιαίου οπτικού μηχανισμού, προξενεί περαιτέρω άχθος, κάτι που για τα μικρότερα ιδρύματα αποτελεί ένα επιπλέον πρόβλημα. Και τέλος, θα ήθελα τα σχόλιά σας για το σχόλιο του Ολλανδού κυβερνήτη του Ολλανδού διοικητή συμμετέχοντας στο Συμβούλιο ότι δεν είναι αποτελεσματικός ο εποπτικός μηχανισμός και τα ποσά που εντοπίζονται ως έλλειψη για τα περισσότερα ιδρύματα. Εάν συμφωνείτε, ποια είναι η αποψή σας για την ε, τοποθέτηση του Ολλανδού διοικητή της Ευρωπαϊκή Κεντρικής Τράπεζας. Regarding methodology μεθοδολογία για την αξιολόγηση του κινδύνου και την ε, αρχή της αναλογικότητας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εφαρμόσουμε την αρχή της αναλογικότητας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κάνουμε μια σωστή διάκριση μεταξύ σημαντικών και λιγότερο σημαντικών ιδρυμάτων. Για τα λιγότερο σημαντικά ιδρύματα, ο βαθμός αναλογικότητας βρίσκεται στα χέρια των εθνικών εποπτών όπως η σύσταση που κάναμε για τα μερίσματα λόγου χάρη. Ήδη εσείς την απευθύνατε στα μεγαλύτερα ιδρύματα και απεστάλλει τους εθνικούς επόπτες ώστε να την υλοποιήσουν αναλογικώς, βάσει της αρχής αναλογικότητας, όπως το θεωρούσαν δέον, στα λιγότερα σημαντικά ιδρύματα. Για αυτήν την κατηγορία λοιπόν δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η αρχή της αναλογικότητας εφαρμόζεται σωστά. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να λάβουμε υπόψη ενός το δυνατόν καλύτερα τις διαφορές μεταξύ σημαντικών ιδρυμάτων. Κάποια είναι πολύ μεγάλα, με πολύ προηγμένα μέσα, όπως ε, τα εννέα μεγαλύτερα ιδρύματα εντός των 23 μεγάλων τραπεζικών ομίλων, και μετά υπάρχουν κάποια τα οποία είναι μεγάλα σε σχέση με τις διαστάσεις των κρατών τους. Μπορείτε να μας ενημερώσετε γι' αυτό, για την υλοποίηση της αρχής της αναλογικότητας ή να μας ενημερώνετε εδώ στο Κοινοβούλιο συστηματικά. Θα ήθελα μια γραπτή δήλωση, διότι λαμβάνω πολλές ερωτήσεις και κάποια ζητήματα τα θίξατε κι εσεί οι ίδια προς στιγμή. Ως την αξιολόγηση κινδύνου στο ΣΡΕΠ να τονίσω ότι εξοπλίζουμε πλήρως το πλαίσιο της Τραπεζικής Ένωσης. Δεν είναι κάτι που έχουμε επινοήσει στον εποπτικό μηχανισμό. Ως προς το ανακρέντιτ. Την αναλυτική βάση δεδομένων οι λεπτομερέστατες πληροφορίες που θέλουμε συχνά απαντώνται, τις βρίσκουμε. Οι επόπτες των μικρότερων τραπεζών είναι μάλιστα αυτοί που πιο πολύ ενδιαφέρονται να δώσουν τόσο λεπτομερείς πληροφορίες. Διότι ακριβώς αφορούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι σημαντικότατες για την οικονομία. Αυτός είναι ο λόγος που υπάρχουν τόσο λεπτομερείς Πληροφορίε βεβαίω υπάρχει στενός συσχετισμό μεταξύ του λεπτομερού χαρακτήρα και τη πρόκληση επιπλέον άχθου. Υπήρχε μια συγκριτική ανάλυση κόστου από τι εθνικέ αρχέ τι εθνικέ κεντρικές τράπεζε όταν αποφασίστηκε. Θεωρήθηκε ότι δεν ήταν επαρκή αλλά θα περιμένουμε και τις αντιδράσεις των Ιδρυμάτων των χωρών. που θεώρησαν ότι δεν αρκούν. Όσο για το κατά πόσο είναι αποτελεσματικά όλα αυτά, να σου δώσω ένα παράδειγμα. Είναι δύσκολη δουλειά μας, είναι περίπλοκη. όπως με την μη μεταφορά της οδηγίας για την εξυγίανση και τη διάσωση. Οι εθνικοί επόπτες πρέπει να ξέρουν το νομικό πλαίσιο εντός του οποίου πρέπει να λειτουργούν. Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα πρέπει να γνωρίζουν και άλλα 19 εθνικά πλαίσια. Επειδή όμως ε, οι αποφάσεις καθυστερούν κατά αυτόν τον τρόπο, να πω το εξή. Ε, είναι η πρώτη χρονιά. Τα πάντα για μας είναι καινούρια μέχρι τον Νοέμβριο του 2015. Οπότε πρέπει να έχουμε συγκεκριμένες ε, συγκεκριμένε πολιτικέ κατευθύνσει για να πάρουμε τι σωστέ αποφάσει, όσο δυνατόν περισσότερο, αλλά χρειαζόμαστε λίγο χρόνο, δεν πρέπει να βιαστούμε, για να μην ληφθούν αποφάσει που θα, ήταν, θα δημιουργούσαν κακό προηγούμενο. Αυτό βέβαια είναι ένα πρόβλημα που ελπίζουμε ότι θα λυθεί μετά το πρώτο δωδεκάμινο λειτουργία. Κατά τα άλλα, ορισμένα χρονικά πλαίσια ορισμένες προθεσμίες που είχαν ήδη προβλεφθεί από εθνικούς επόπτες είναι δύσκολο να τηρηθούν και δεν έχουν ε, πολύ μεγάλη σχέση με την πραγματικότητα. Δηλαδή για να επακούσει κανεί και στου κανόνε του κοινοποπτικού μηχανισμού τα πράγματα γίνονται λιγότερο εφικτά και ακόμη και αν πρέπει να λάβει υπόψη και την ε, τραπεζική αρχή, ε, τα πράγματα εμπλέκονται ακόμη περισσότερο. Το ίδιο και με του πολύ μεγάλου ομίλου. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι απλοποιούμε, απλουστεύουμε κάπως τη διαδικασία σε αυτές τις περιπτώσεις. Νομίζω ότι έχουμε εξαιρετικού συνεργάτες που εργάζονται όσο πιο σκληρά μπορούν για να φέρουν αποτελέσματα στο δυνατόν πιο γρήγορα. Συνήθω βλέπουμε ένα προσχέδιο τη απόφαση ε, για την οποία πρέπει να λάβουμε αμέσω απόφαση και τελευταία στιγμή και πολλέ φορέ και καθυστερημένα. Δεν είναι πολύ εύκολο λοιπόν πάντοτε να είμαστε βέβαιοι ε, να σας πω ότι ούτως ή άλλως θα έχουμε ένα εργαστήριο για την EBA και την, αρχή, την εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας στο πλαίσιο του ε, θεσμικού πλαισίου την επόμενη εβδομάδα, την Παρασκευή. Επόμενος ομιλητής ο κύριος Τζάνι. Ο κύριος Σίμων αν ήθελε να αναλάβει την Προεδρία για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ. Έχω τρεις ερωτήσεις. Η πρώτη αφορά τα επόμενα τεστ κόπωσης. Σε μια πρόσφατη συνέντευξη δηλώσατε ότι δεν θα γίνουν το 2015 τεστ κόπωσης αλλά το 2016. Η ερώτησή μου είναι εάν θα αλλάξουν τα κριτήρια για την ανάλυση και πιο συγκεκριμένα, εάν σκοπεύετε, τον κίνδυνο έκθεση στα παράγωγα να τον θεωρήσετε κεντρική σημασία για ισολογισμού ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων κατά κύριο λόγο. Η δεύτερη ερώτηση αφορά την ε, περίπτωση της ETA Bank και την εφαρμογή της οδηγίας για την εξυγέννηση και τη διάσωση. Τις δυσκολίες του γερμανικού και αυστριακού τραπεζικού συστήματος χωρίς ε, αρχές εγγύησης, πώς την αξιολογείτε, πώς θα προχωρήσετε με την υλοποίηση της νέας οδηγίας. Και πώς αξιολογείται τον ενδεχόμενο κίνδυνο πτώχευσης ε, και τις επιπτώσεις στο γενικότερο γερμανικό και τραπέζικο ε, σύστημα. Και επίσης μια ερώτηση για την τράπεζα την ε, Monte de Paschi της Σιένα, η οποία βρέθηκε σχεδόν σε κατάσταση πτώχευσης, αλλά με αύξηση 3 δις ευρώ που έγινε πρόσφατα. Θέλω να ξέρω με την αύξηση αυτού του κεφαλαίου η τράπεζα ξαναπέρασε στους συντελεστές του σωστού κεφαλαίου που απαιτούνται και αν η κατάσταση θεωρείται ότι ξομαλύνθηκε ή αν θα απαιτήσετε περαιτέρω βήματα για να εξομαλυνθεί, να εξηγενθεί τελείως κατάσταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σε ό,τι αφορά τα τεστ κόπωση, όντω πρέπει να γίνει πολλή δουλειά. Είναι πολύ δύσκολο για 133 τραπεζικού ομίλου να γίνονται τέτοια τεστ. Και εάν γινόταν μια τέτοια διαδικασία κοινή το 2015, θα πρέπει ήδη να έχουμε ξεκινήσει. Ταυτόχρονα με την εποπτεία θα ήταν υπερβολικό ο Ούτε οι ΗΠΑ δεν κάνουν αυτό το πράγμα δύο φορές ε, μέσα σε ένα χρόνο. Αλλά θα συμμετάσχουμε στα τεστ της ε, EBA το 2016 όπως έχουν προγραμματιστεί. Έχουμε αρχίσει να σκεφτόμαστε το πώς θα γίνει σωστή κατανομή αλλά η πραγματική δουλειά για το 2016 έτσι κι αλλιώς ξεκινάει από το Σεπτέμβριο φέτος ως προς την έλλειψη μεταφοράς της οδηγίας για τη διάσωση και την ε, εξυγίανση. Η κατάσταση είναι αρκετά σαφής. Είτε έχει μεταφερθεί είτε όχι. Εάν όχι, πρέπει να δούμε την κατάσταση στην ε, κάθε μια χώρα που δεν έχει κάνει τη μεταφορά. Υπάρχουν εθνικοί κανόνες για τη διάσωση, Οπότε πρέπει να γνωρίζουμε καλά τους νόμους για να μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε αποτελεσματικά. Εάν δεν υπάρχουν τέτοιοι νόμοι, αν δεν υπάρχει σχετική νομοθεσία, έρχομαστε σε επαφή με τα Υπουργεία Οικονομικών. Όπως και η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει κάποια μορφή συνεργασία με τις ε, Ιωνίοι Εποπτικές Αρχές πριν δημιουργηθεί το πλαίσιο εποπτείας. Ξέρουμε λοιπόν ποια είναι η κατάσταση σε ένα χώρα και θέλουμε να υπάρξει πλήρης μεταφορά της οδηγίας. Διότι η δουλειά μας δεν είναι ότι καθίσταται αδύνατη, γίνεται απλώς πολύ πιο περίπλοκη. Με ρωτήσατε για την Μοντεπάσκη. Κοιτάξτε, η Μοντεπάσκη είχε πρόβλημα κεφαλίου, έπρεπε να το καλύψει έκανα την απαραίτητη κίνηση πριν τις 26 Ιουλίου που ήταν η προθεσμία και νομίζω ότι η κίνηση ήταν θετική. Δεν έχω όμως πολλά να προσθέσω. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μονό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, ανακοινώσατε αρχές Ιουνίου ότι θα κάνετε καινούργιες δοκιμές κόπωσης για 123 συστημικές τράπεζες. Πρώτο ερώτημα. Με ποια μέθοδο θα γίνουν αυτές οι δοκιμές. Πέρυσι είχατε πει ότι οι δοκιμές που κάνατε μετρούσαν τις επιπτώσεις ενός σενάριου κρίσης αλλά ότι δεν είχαν συνδυαστεί τώρα που υπάρχει και ο αποπληθωρισμός η ΕΚΤ έχει προετοιμαστεί για αυτή την αντιμετώπιση του κινδύνου του αποπληθωρισμού επίσης για τα επιπτώσεις της κρίσης στις συστημικές τράπεζες τι θα κάνετε και πώς θα αντιμετωπιστεί μια πιθανή ένοπλη σύραξη. Επίσης μίλησε ένας συνάδελφος για την κατάσταση με τα CDS και για μένα και εγώ πιστεύω ότι έχουν υποτιμηθεί σε περίπτωση μίζωνος κρίσης η φεργιότητα των τραπεζών δεν θα απειληθεί. Τέλος, θεωρείτε ότι είστε αρκετά ανεξάρτητοι σε αυτήν τη δουλειά εποπτείας που κάνετε ως προς το opting της ΕΚΤ. Euh, euh, Ευχαριστώ για την μέθοδο των ε, δοκιμών κοπόσεως πέρυσι ή μάλλον για το 2016 θα τα κάνουμε με την EBA, EBA αλλά ακόμα δεν τα έχουμε αρχίσει τη συζήτηση. Το φινόπωρο. Όσο για τα σενάρια, πολλοί παράγοντες παρεμβαίνουν στα σενάρια αυτά. Η Κομισιόν καταρχήν. Το SRB, το Συμβούλιο δηλαδή Συστημικού Κινδύνου, παίζει σημαντικό ρόλο και άλλα τμήματα της ΕΚΤ για, που ασχολούνται με την χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Τελικά όμως η ΕΜΠΑ, το EBA αποτιμάει τα σενάρια και τις δοκιμές. Είμαστε και εμείς μέλος της EBA αλλά δεν, πιστε, δεν ψηφίζουμε. Τα μέλη ψηφίζουν άμεσα. Όλα αυτά λοιπόν θα γίνουν με συνεργασία και συνδυασμό και στο τέλος το ΚΕΜ, το SSM, θα βγάλει τα συμπεράσματα των αποτελεσμάτων της EBA. Έτσι αποφεύγονται οι διαμάχες και τα αντικρουόμενα συμφέροντα. Γιατί θα έχουν συνεργαστεί όλοι οι αρμοδιότεροι παράγοντες. Μιλήσατε και για συνδυασμένα σενάρια που δεν τα εξετάζουμε εμείς από τις δοκιμές. Αυτή είναι ακριβώς η διαφορά. Μιλάμε τώρα για στρες κόπωσης, για δοκιμές κόπωσης σε μεγάλη κλίμακα. Υπάρχουν όμως και άλλα προγράμματα και ασκήσεις μικρότερης κλίμακας που δεν γίνονται πολύ συχνά αλλά τακτικά πάντως. Κάθε φορά που ένας επόπτης, ας πούμε αν εγώ θέσω ένα ερώτημα στην ομάδα μου. Τι θα γινόταν εάν και μετά δώσω μερικά στοιχεία για να μου πούν τι επιπτώσεις θα είχε η υπόθεση που κάνω. Και αυτό τι είναι, τι άλλο είναι. Είναι δοκιμή κοπόσεως και αυτό. Συνδυασμός δηλαδή διαφόρων υποθετικών παραγόντων. Είναι και αυτό λοιπόν μέρος της τρέχουσας δουλειάς του επόπτη να κάνει τέτοιου είδους συγκεκριμένα stress test. Όταν αφορά βέβαια μικρές λιανικές τράπεζες ή τεράστιες και πολύπλοκες τράπεζες είναι αλλιώς τα πράγματα, όπως τα CDS, αλλά όλα αυτά λαμβάνονται υπόψη. Μπορούσαμε να πούμε ότι ξεχάσαμε να δοκιμάσουμε τον α ή τον β παράγοντα κινδύνου, αλλά δεν είμαι βέβαιη ότι ξεχνάμε, γιατί κάνουμε πάρα πολλές δοκιμές και τα σκεφτόμαστε όλα λεπτομερώς τις επιπτώσεις ορισμένων καταστάσεων και γεγονότων. Τώρα αν αισθάνομαι ελεύθερη και ανεξάρτητη είναι φυσικά, απολύτως. Και είμαι γνώμων προς την ΕΚΤ που μου χορηγεί ένα πλαίσιο και τα μέσα για την, και στήριξη για την άσκηση των καθηκόντων αυτών ώστε να αφιερώνομαι αποκλειστικά στην εποπτεία τα υπόλοιπα τις μισθοδοσίες, τις προσλήψεις, τη διοντολογία κτλ. Αυτά μας τα δίνει η ΕΚΤ έτοιμα και αυτό είναι πολύ καλό για να αφιερωνόμαστε αποκλειστικά στη δουλειά μας ανεξάρτητα και το ότι επελέγει από το Κοινοβούλιο για αυτή τη θέση είναι μια πρόσθετη εγγύηση ανεξαρτησίας. Αλέν Λαμασούρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, μας είπατε ότι διαπιστώσατε ότι μεταξύ των μελών της Ευρωζώνης υπάρχουν διαφορετικοί εθνικοί κανόνες άλλοι παλαιοί, άλλοι προέρχονται από την εφαρμογή εθνικών επιλογών και ένας από τους ρόλους σας είναι να δημιουργείτε κάποια σύγκληση για να μην είναι αντιφατικοί αυτοί οι κανόνες. Μπορείτε να μας πείτε όμως μήπως αυτή τη στιγμή επί ποιων σημείων σημειώνονται σημαντικές διαφορές και ποιες διαφορές υπάρχει ο κίνδυνος να παραμείνουν ακόμη και όταν θα έχει περάσει η μεταβατική περίοδος στην οποία διαπιστώνουμε αυτή τη στιγμή, στην οποία ζούμε αυτή τη στιγμή. Πράγματι υπάρχουν ορισμένες επιλογές εθνικές που προβλέπουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες και από τον Νοέμβριο του 2014 οι επιλογές που είναι στα χέρια των εποπτών δηλαδή τα δύο τρίτα περίπου το ΚΕΜ έχει το καθήκον και την υποχρέωση να αποφασίσει, να δει ποιες θα κρατήσει από αυτές τις επιλογές. Τώρα το μελετούμε, θα θέλαμε βέβαια την μέγιστη δυνατή εναρμόνιση, αλλά να γίνει αυτή και με αυστηρά κριτήρια. Έχουμε μια ομάδα εργασίας που θα διατυπώσει προτάσεις και πρέπει να σας πω ότι με έχει ενθαρρύνει πολύ και ευχάριστα εκπλήξει η θέληση που επιδείχτηκε για να γίνει αυτή η προσπάθεια. Οι περισσότεροι ρες από αυτές τις εθνικές επιλογές θα εναρμονιστούν με αυστηρό τρόπο, ακριβέστατο τρόπο ε, μερικές βέβαια μπορεί να απορρέουν από συμφωνίες όπως τον Δανέζικο Συμβιβασμό, ασφαλιστικές εταιρείες, το καθεστώς των αγγλικού δικαίου ορισμένων δανείων που προκύπτουν, που θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικά κέρδη που μπορεί να συνεχίζουν να εμφαίνονται στο ενεργητικό των τραπεζών. Υπάρχει λοιπόν εκεί μεγάλη ευχέρεια ελιγμών και διαφορετικές καταστάσεις διαφορετικών τραπεζών. Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα, καμιά δεκαριά πιο δύσκολες περιπτώσεις. Κάναμε μία μελέτη αξιολόγηση, τα αποτελέσματα θα τα έχουμε τις επόμενες μέρες και κάθε φορά που υπάρχει σημαντική επίπτωση θα λάβουμε υπόψη μας τα νόμιμα συμφέροντα ή προσδοκίες, θεμητές προσδοκίες των τραπεζών που προκύπτουν από αυτές τις εθνικές επιλογές για να είμαστε λίγο πιο ευλίγιστοι, ευέλικτοι και λιγότερο αυστηροί με στόχο πάντα να καταλήξουμε σε μία σύγκληση ώστε οι επιλογές αυτές στο βαθμό που είναι δυνατόν να τύχουν εναρμόνισης δεν ξέρω όμως ποια θα είναι η τελική επίπτωση και η τελική απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου. Αλλά μέχρι τώρα η ποιότητα των συζητήσεων ήταν θα ενθαρρυντική. Στο και το Κοινοβούλιο ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για αυτή την ε, μελέτη αντικτύπου στην οποία αναφερθήκατε. Πέτρα Ζήμων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ανουή, για την παρουσίασή σας και για αυτά που είπατε για τις ερωτήσεις του κυρίου Γκίγκολ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το ανακρεντήτ. Και θέλω να συνεχίσω ε, σε αυτή την ε, γραμμή σκέψης. Από ό,τι ακούω από τις μικρότερες τράπεζες για παράδειγμα, ότι παρά το ότι προσαρμόστηκαν αυτά που τους ζητούνται στο ανακρεντήτ, βγήκαν δηλαδή ορισμένα που δεν είχαν έννοια από πρώτη μεριά, αλλά παρόλη αυτή την αλλαγή πρέπει για αυτές τις πιστώσεις ε, των 25.000 ευρώ 150 στοιχεία του ζητάνε. Για παράδειγμα για την βελτίωση ενός μικρού γκαράζ. 150. Απίστευτος αριθμός. Πώς είναι δυνατόν. Θεωρείτε ότι χρειάζεστε όλα αυτά τα στοιχεία. 150 κουτιά πρέπει να συμπληρώσουν. Έγινε καμία δημόσια διαβούλευση γι' αυτό. Υπήρχε καμία διαδικασία που να μας επιτρέπει να καταλάβουμε πώς είναι δυνατόν χρειάζεται τόσα στοιχεία. Σας παρακαλώ είτε σήμερα ή ίσως μετά γραπτός ή θα σας ήμουν επίσης πιο ευγνώμων αν μπορείτε σε μια περαιτέρω συνάντησή μας εδώ στην Επιτροπή να μας εξηγήσετε γιατί πώς είναι δυνατόν να δικαιολογούνται τόσα στοιχεία που σημαίνουν ε, πολύ γραφειοκρατικό κόστος και κόστος. Δεύτερον, επικοινωνία με τις τράπεζες. Έχω μία επιστολή τώρα της τράπεζας, ε, ε, μιας μικρής συνεργατικής τράπεζας από την Ρινανία Βεσφαλία Παλατινάτο. Και εκεί μας λένε πόσα πρέπει να πληρώσουν στην ΕΚΟΥΤΟΥ με βάση την απόφαση 207 του 2015. Πρέπει λοιπόν οι συνεργατικές τράπεζες να στείλουν στοιχεία πώς θα πρέπει να σταλούν τα στοιχεία και πώς θα τα ε, πλαισιώσουν πρέπει να σταλούν στα αγγλικά και με μία μη επίσημη ε, ε, τώρα τα λέει ανάποδα ο μιλητής πρέπει να σταλούν στα γερμανικά με μη επίσημη αγγλική μετάφραση τι σημαίνει αυτό τους επιτηρείτε άμεσα ή άμεσα μέσω της εθνικής, ε, μέσω της εθνικής εποπτικής αρχής. Δεν είναι δυνατόν όλα τα στοιχεία να στέλνονται μόνο μέσω της εθνικής γλώσσας και να υπάρχει επίσημη μετάφραση. Και σε τι πλαίσιο μπορείτε να εγγυηθείτε ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Ε, Ευχαριστώ. Όσον αφορά το Anna Credit. Επιβεβαιώνω αυτό που είπα και πριν. το επίπεδο αναλυτικών πληροφοριών, το επίπεδο λεπτομέρειας, είδαμε ότι είχε αποφασιστεί πριν αναλάβουμε τα εποπτικά μας καθήκοντα. Έγινε μία ανάλυση του υπέρ και του κατά, του κόστους ωφέλους. Έγινε όμως από τις ε, εθνικές κεντρικές τράπεζες, όχι κατά ανάγκη από τους ε, εθνικούς επόπτες γιατί ήταν ένα πρόγραμμα που είχαν ξεκινήσει οι κεντρικές τράπεζες πριν αρχίσει να λειτουργεί το SSM. Επίσης, γιατί αυτή η διαδικασία δεν προβλέπει περαιτέρω δημόσια διαβούλευση σε αυτή τη βάση. Αυτή τη στιγμή προετοιμάζουμε μία αναλυτική ιστοσελίδα του Anacredit για να έχουμε μία γραμμή επικοινωνίας με τους φορείς που εμπλέκονται στο Anacredit για να συνοηθούμε για το πώς θα προχωρήσουμε και να ζητήσουμε και από την ευρύτερη κοινή γνώμη συμβουλές, δηλαδή από τις τράπεζες που θα στέλνουν στοιχεία για το ανακρέντιτ και για να βοηθήσουμε μέσω, ξέρετε, αυτού του λεγόμενου FAQ, ε, συνήθεις ερωτήσεις. Στέλνουμε λοιπόν και στους εθνικούς επόπτες και στις τράπεζες το μήνυμα να αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα, αυτή την ιστοσελίδα για να μας απαντήσουν. Τώρα για το Εποπτικό Συμβούλιο, το SRB. Υπάρχουν ε, διαφορές απόψεων για ποιο επίπεδο λεπτομέρειας χρειάζεται. Αλλά ορισμένες χώρες, ορισμένες εποπτικές αρχές και από ό,τι φαίνεται και ορισμένες τράπεζες, πραγματικά επιμένουν ιδιαίτερα στα αιτήματά τους για πολλές λεπτομέρειες. Πρέπει λοιπόν όλοι οι ενδιαφερόμενοι να ληφθούν υπόψη. Και ορισμένοι έχουν πολύ ε, κατηγορηματικές απόψεις. Και η Κεντρική Τράπεζα οπωσδήποτε θα τα λάβει υπόψη της. Καταλαβαίνω ότι θα θέλατε να σας πω κάτι πιο σαφές. Αλλά δεν είναι κάτι που το ξεκινήσαμε εμείς δεν είναι κάτι που το διαχειρίζουμε. Τώρα όσον αφορά τις μεταφράσεις, ε, ναι, το γλωσσικό θέμα στην Ευρώπη είναι περίπλοκο. Μάλλον πιο περίπλοκο από ό,τι περιμέναμε. Και έχω ζητήσει περισσότερο προσωπικό. Αλλά το τμήμα ΕΚΟΥΤΟΥ του SSM και το εθνικό τμήμα του SSM προσπαθούν να συνοηθούν για να δουν ποιος θα κάνει τι όσον αφορά τις μεταφράσεις. Τι θα πρέπει να μας δώσουν οι εθνικοί επόπτες και τι η κεντρική τράπεζα, η ΕΚΤ. Κάνουμε πολλές μεταφράσεις, ξέρετε, πολλές. Αλλά εάν κάτι δεν γίνεται, ε, πείτε μας, πείτε μας. Πείτε μας τι λείπει, τι πρέπει να κάνουμε και θα δούμε εάν είναι αρμοδιότητα των εθνικών εποπτών στο SSM ή της ε, ΕΚΤ στο SSM. Τώρα, τη σχέση που έχει η ΕΚΤ με τις εθνικές τράπεζες που θέλουν να συντάσσουν τα κείμενά τους ε, στην ε, δική τους γλώσσα, ξέρετε είμαι ιδιαίτερα βαριά, είμαι ιδιαίτερα απαιτητική, ακόμη και στα email, ακόμη και στα παραρτήματα των email, τα συνημένα, επειδή όλα αυτά είναι λίγο λιγότερο επίσημα, μπορεί να υπάρχει κάποια τάση ε, για κάποια ε, χαλαρότητα όσον αφορά τη χρήση της εθνικής γλώσσας. Αλλά εγώ επιμένω και πείτε μας τι θα έπρεπε να έχει μεταφραστεί και δεν έχει μεταφραστεί και θα περάσω το μήνυμά σας. Hawkmark Σας ευχαριστώ Πολλές από τις ερωτήσεις προς εσάς έχουν να κάνουν με το τι πρέπει να αλλάξει και τι όχι και πώς πρέπει να ασχοληθούμε με τις νέες ευκαιρίες. Όμως ενδιαφέρον θα είχε να ακούσουμε από εσά όχι μόνο πόσο είναι μισοάδιο το ποτήρι αλλά και πόσο είναι μισογεμάτο. Εάν δείτε τον Ευρωπαϊκό Τραπεζικό τομέα σήμερα με νέα νομοθεσία για τις κεφαλικές απαιτήσει την διάσωση και εξυγίανση και πολύ πιο εναρμονισμένη υποπτία. Πώς θα περιγράφατε την κατάσταση, έστω τις αδυναμίες από τη δική σας την οπτική γωνία της Ευρωπαϊ... του Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Κλάδου. Ποιες είναι οι αδυναμίες, πέρα από το γεγονός ότι κάποια κράτη πρέπει να εφαρμόσουν πλήρως την νομοθεσία. Σε τι, ε, ε, ε, τι έχει αλλάξει σήμερα σε σχέση με το τι συνέβαινε πριν από πέντε χρόνια. Ποιε είναι οι συγκεκριμένε σημερινέ αδυναμίε που να επιληθούν. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα, για να δούμε και το υγιέ στοιχείο στι τράπεζε Ό,τι αφορά τον κανονισμό, έχει γίνει μεγάλη πρόοδο. Καλύτερη νομοθεσία των τραπεζών, άντληση διδαγμάτων από την κρίση, μέρος των δυσκολιών είναι ότι βρισκόμαστε σε μετάβαση με, το, ε, με την οδηγία για τις Πολιτικές απαιτήσει, τέσσερα με, την, ε, με τον κανονισμό για την εξυγίανση και την διάσωση. Είναι πολλοί κανόνες. Υπάρχει και η καλύτερη νομοθεσία, το Better Regulation. Πρέπει λοιπόν να ε, ξέρουμε ότι θα μας πάρει ακόμα κάποιους μήνες ή χρόνια μέχρι όλα αυτά να λάβουν σάρκα και Σε ό,τι αφορά τον τραπεζικό κλάδο Όλες οι τράπεζες της Ευρωζώνης έχουν, καταβάλει έχουν καταφέρει πρόοδο ενισχύοντας τους ισολογισμούς τους. Και μάλιστα σε ένα περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις. Παρά τις προσπάθειες όμως να ενισχυθούν οι θέσεις ε, στο προς τα κεφάλαια τα τελευταία χρόνια, οι τράπεζες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ε, δυσκολίες, τουλάχιστον σε δύο μέτωπα. Πρώτα απ' όλα οι τράπεζες της Ευρωζώνης συνεχίζουν ε, να γνωρίζουν αναταράξεις λόγω της χαμηλής κερδοφορίας που συνδυάζεται με κυκλικά και διαρθωτικά αδιέξοδα. Ε, οι κυκλικές αδυναμίες έχουν να κάνουν από την ε, ισχνή οικονομική ανάκαμψη και πέρα από τις κυκλικές εξελίξεις, ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει τις τράπεζες είναι η ταχύτητα με την οποία προσαρμόζουν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα στην νέα πραγματικότητα. Αυτήν που προκύπτει λόγω των ρυθμιστικών απαιτήσεων. Μια δεύτερη μεγάλη πρόκληση που πιέζει πολύ τις τράπεζες στις πλέον ευάλωτες χώρες έχει να κάνει με τα προβληματικά στοιχεία του ενεργητικού ή τα ενδυνάμει προβληματικά στοιχεία του ενεργητικού και τις ε, δυνατότητες δανειοδότησης των τραπεζών. Για τα προβλήματα με τα μη κερδοφόρα δάνεια αυτό απαιτεί αλλαγή συνολικά της προσέγγισης παρόλο που δεν υπάρχει μία λύση ίδια για όλους. One size. Πρέπει να δούμε τις κακές τραπεζικές πρακτικές, τις οικονομικές ε, συνθήκες που δεν είναι καλές, την ε, δυσκολία πρόσθεσης στην ανάκαμψη, την ε, δυσκολία προσαρμογής στα συστήματα, πράγματα που ξεπερνούν όμως την εντολή και τις αρμοδιότητες του υποπτικού μηχανισμού. Συνολικά η χαμηλή κερδοφορία με ε, στοιχεία των ενεργητικού που έχουν κληροδοτηθεί από το παρελθόν και δεν δίνουν μεγάλες επιστροφές, δεν επιτρέπει να δημιουργηθούν οι σωστές ασπίδες των κεφαλαίων εντό εισαγωγικών για να αντιμετωπιστούν οι κραδασμοί της ε, οικονομίας γενικότερα. Πάντως πρόοδος ε, έχει καταβληθεί σε κάποια πράγματα μέχρι να φτάσουμε σε πιο οριστικές βελτιώσεις. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Καλά νέα αυτά. Ο κύριος Μαυρίδης. Thank you, Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τρεις πολύ σύντομες ερωτήσεις. οι οποίες είναι αλληλένδετες. Και έχουν να κάνουν περισσότερο με τα οικονομικά παρά με τα λογιστικά το να χρησιμοποιούμε μαθοποιημένα στοιχεία μπορεί να ε, αποκρύπτει συγκεκριμένα προβλήματα για συγκεκριμένες χώρες. Στην περίπτωση της Κύπρου, πάνω από 50% των χαρτοφυλακίων, των δανείων ε, στα στοιχεία του ενεργητικού θεωρείται ότι δεν αποδίδουν. Ωστόσο, ταυτόχρονα οι τράπεζες στην Κύπρο φαίνεται να έχουν κερδοφορία. Ήθελα λοιπόν από οικονομική σκοπιά μια απάντηση. Και η δεύτερη σύντομη ερώτησή μου. Οι ελληνικές τράπεζες ε, που λειτουργούν στην Κύπρο, βλέπετε να υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε αυτό. Εάν υπάρξει πτώχευση στην Ελλάδα με το κρατικό χρέος, ε, έχετε προβλέψει τίποτα μέτρα. Και τρίτη σύντομη ερώτηση. Όπως δηλώσατε, στην αρχική τοποθέτηση συμφωνία σε πολιτικό επίπεδο για την Ελλάδα θα ήταν ικανοποιητική. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι η εξή. Πιστεύετε ότι η παράταση του προγράμματος θα έπαβε την ε, εκροή κεφαλαίων και των καταθέσεων από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Ευχαριστώ. Σύντομες ερωτήσεις αλλά δύσκολες. χρήση δεδομένων που δεν καλύπτουν απαραίτητο συγκεκριμένα προβλήματα σε συγκεκριμένε χώρε ή που τα αποκρυπτούν. Τα δεδομένα είναι ένα πρώτο σημείο αφετηρία. Όμω είναι σημαντική και η κρίση, η δυνατότητα των εποπτών να κρίνουν. Χρειαζόμαστε όμω ενός είδου θερμόμετρο, μία καταγραφή τη θερμοκρασία και μετά προχωρούμε σε αποτίμηση. Σε ό,τι αφορά τη σχέση των στοιχείων έκθεσης που ε, δεν αποδίδουν και το κέρδος, στην κερδοφορία, ε, το συνδετικό στοιχείο μεταξύ των δύο είναι η κάλυψη. Το κατά πόσον καλύπτονται δηλαδή αυτές οι περιπτώσεις έκθεσης ε, που δεν αποδίδουν. Για το θέμα αυτό όπως και για άλλα, προσπαθούμε να ακολουθήσουμε τις βέλτιστες αποπτικές πρακτικές. Χρειαζόμαστε ε, να ακολουθήσουμε πρακτικές όπως αυτές της Ιρλανδίας σε αυτή την περίπτωση, όπου ήταν αποτελεσματικές οι κινήσεις τους. Θα δούμε μήπως αυτό αποδίδει και σε άλλες ε, χώρες μαζί με την ε, εφαρμογή των όσων προβλέπει ο εποπτικός μηχανισμός. Σε ό,τι αφορά τις συνέπειες για την Κύπρο, και ιδίω αν κάτι συμβεί με τι ελληνικέ τράπεζε. Πρέπει να πω ότι ο ενιαίο οπτικό μηχανισμό διευκόλυνε πολύ σε αυτό το πλαίσιο και για την Κύπρο και για την Ελλάδα. θα επιτρέψει και στην Ελλάδα και στην Κύπρο να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα επικοδομητικά. Όπως ξέρετε, οι φυγατρικές ελληνικών τραπεζών στην Κύπρο, ε, στην Κύπρο έχουν ενισχυθεί σωστά ε, στα κεφαλαία τους. Ε, δόθηκαν ποσά από τις ομίλου τους. Δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Και όπως λέμε στη δική μας τη διάλεκτο, είναι και φερέγγιες και με ρευστότητα και σε σταθερή βάση. ως προς το πολιτικό επίπεδο. Κοιτάξτε, δεν είμαι πυρηνική φυσικός, είμαι απλός υπόπτης. Αποτιμούμε τις καταστάσεις, τον κίνδυνο και μετά σχεδιάζουμε κάποιες ενέργειες ε, βάσει του νομικού πλησίου. Ελπίζω ότι αυτό απαντά στην ερώτησή σας. Πρόεδρος. Ο κύριος Μούρεζαν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κυρία πρόεδρε, δύο σύντομα ερωτήματα για δύο τάσεις που παρατηρούμε στο τραπεζικό τομέα. Πρώτον, αυξημένη έκθεση των τραπεζών σε στα δημόσια χρέη. Ερωτώ λοιπόν, το ΚΕΜ έχει αποτιμήσει το ρίσκο που αντιμετωπίζει αυτή η έκθεση στα δημόσια χρέη και αυτό βέβαια οφείλεται και στον μηδενικό κίνδυνο που έχετε αποτιμήσει για ορισμένα δημόσια χρέη. Σε τι ποσοστό μπορεί μια τράπεζα να κρατήσει δημόσια χρέη ή να αγοράσει με τρόπο όμως που να μην διαταράξει τον τραπεζικό τομέα και την οικονομική δραστηριότητα στην Ευρώπη. Δεύτερο ερώτημα. Έκθεση των ισολογισμών των μεγάλων τραπεζών. Πράγμα που παρατηρήθηκε στην πρώτη φάση της κρίσης. Ερωτώ λοιπόν, έχετε καμία συγκεκριμένη άποψη για την έλλειψη για τις εκτός ισολογισμού εκθέσεις ως τρόπο για να καλύψουμε την έλλειψη κεφαλαίων. Σας παρακαλώ να μην μιλάτε εδώ μέσα. Μεταξύ σας. Ευχαριστώ για τους κινδύνους με τα δημόσια χρέη. Ε, ήδη είπα ότι μαθαίνουμε κατά τη διάρκεια της κρίσης σιγά σιγά ότι η έκθεση δημόσιου χρέους δεν είναι κίνδυνος για τα πεπραγμένα της τράπεζας ή θα έπρεπε να υπάρχει και βέβαια και κάποιο όριο στην έκθεση αυτή. Αρχίσαμε να το αναλύουμε αυτό και από την Επιτροπή της Βασιλείας. Ελπίζουμε να δημιουργηθεί κάποιο διεθνές πρότυπο γιατί καλύτερο είναι να υπάρχουν διεθνείς κανόνες που να μπορούν να εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ευρώπη ή και στην Ευρώπη. Θα δούμε λοιπόν ποια θα είναι τα συμπεράσματα. Θα χρειαστεί πάντως κάποια προοδευτική εφαρμογή των νέων κανόνων για να μην δημιουργηθούν προβλήματα με κάποια πιο απότομη αλλαγή. Αλλά συχνά το λέμε ότι υπάρχει κάποιος κίνδυνος για και πρέπει να ληφθούν υπόψη κανόνες διαφοροποίησης ώστε προοδευτικά να αρχίσουμε να κινούμαστε προς βελτίωση της κατάστασης χωρίς να περιμένουμε τους τελειωτικούς κανόνες. Τώρα για τα εκτός ισολογισμού. Ίσως να μην το είπαμε αρκετά κατά την συνοπτική αξιολόγηση, αλλά κάναμε μία αυστηρή αξιολόγηση αυτών των εκθέσεων όχι μόνο στις δοκιμές αλλά και η συνοπτική αξιολόγηση το εξέτασε αυτό και τα παράγωγα και τη, στη μεθοδολογία της EBA λήφθη αυτό υπόψη. Οι τράπεζες που εκτέθηκαν σε τέτοια προβλήματα εξετάστηκαν με έξι σενάρια, δύο από τα χειρότερα των οποίων χρησιμοποιήθηκαν και ως δεδομένα για την ε, δοκιμή κόπωσης. Οι κεφαλαιακές ανάγκες αυξήθηκαν αναλόγως με το πρόβλημα. Το ελέγχουμε λοιπόν και αυτό. Δεν είναι και το πιο πολύπλοκο τμήμα της δουλειάς μου προς το παρόν. Ευχαριστούμε πολύ. Βέβαια για τα δημόσια χρέη είναι νομοθετικό το θέμα και το θα το αποφασίσουν οι νομοθέτες, όχι οι επόπτες και οι πέντε πρόεδροι ίσως. Το λένε στην έκθεσή τους. Νίνα Τζιλ. Ευχαριστώ. Πολλά που ήθελα να αναφέρω έχουν ήδη αναφερθεί. Οπότε, έχουμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ κανονισμών και πρόσβασης για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις σε χρηματοδότηση. Γιατί πολλοί στον κλάδο αυτό θεωρούν ότι έχουμε υποβάλει πολλούς κανονισμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα σε σχέση με τις Ηνωμένες Και άρα οι ξένες τράπεζες υπάρχει κίνδυνος να έχουν ε, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ποια είναι η άποψή σας γι' αυτό και σε σχέση με αυτό. Η οικονομία της Ένωσης ε, εξαρτάται περισσότερο από τη χρηματοδότηση από τις τράπεζες σε σχέση και πάλι με τις ΗΠΑ. Βλέπετε να έχει υπάρξει κάποια αλλαγή σε αυτό. Δηλαδή, πώς εξελίσσεται η χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων. Γιατί ανησυχώ επειδή υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές όσον αφορά αυτά που χρειάζονται για παράδειγμα οι μικρομεσαίες στην Γερμανία σε σχέση με την Ισπανία. Και τώρα για το CMU που είναι στο κέντρο της ε, προσοχής μας. Μπορεί να είναι σημαντικό εάν είναι ε, αρκετά λειτουργικό. Έχουμε κάνει ως Κοινοβούλιο μια προσπάθεια να διευκρινίσουμε την κατάσταση και να την κάνουμε πιο διαφανή οι εμπειρογνώμονες θεωρούν θα έπρεπε να υπάρχει ένα μητρό δεδομένων όπου να αναφέρεται κάθε όπου να αναφέρεται κάθε ενέργεια στον τομέα αυτό και να παρακολουθούμε την λειτουργικότητα. Αυτό νομίζει, νομίζετε ότι θα μειώσει τις αμφιβολίες που υπήρχαν για αυτό το εργαλείο, το CMU, στο παρελθόν στην Ευρώπη. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Όσον αφορά τον ε, το κανονιστικό πλαίσιο και τη δυνατότητα χρηματοδότηση τη πραγματική οικονομία, τους καταναλωτές. Δεν νομίζω ότι είναι υπερβολικοί οι κανόνες στην Ευρώπη. Είχαμε πιο χαλαρή εισαγωγή των νέων ρυθμίσεων για το CRD δηλαδή την ε, οδηγία της κεφαλαϊκής απαιτήσεις στις ΗΠΑ ήταν πολύ πιο απότομη και ταχεία η εισαγωγή. Αλλά αυτή είναι τώρα η άλλη όψη του νομίσματος. Επειδή ήμασταν πιο χαλαροί, ορισμένες τράπεζες καθυστερούν ακόμη. δεν αντιμετωπίζουν αρκετά τα μη εξυπηρετούμενα στοιχεία ενεργητικού του παρελθόντος και αυτό σημαίνει πως δεν μπορούν να δανείσουν την πραγματική οικονομία. Η καλά ανακεφαλαιοποιημένες τράπεζες δανείζουν καλά στην πραγματική οικονομία. Οι τράπεζες που δεν έχουν επαρκές κεφάλαιο δανείζουν μόνο σε καλές εποχές. Επειδή βέβαια τότε υπάρχει πολλή δραστηριότητα. Και αυτό δημιουργεί και τις ε, φούσκες. Και όταν προκύψει η κρίση δεν συνεχίζουν να χρηματοδοτούν ή εξαφανίζονται από διάφορους τομείς χρηματοδότησης της οικονομίας και παροχής υπηρεσιών. Δεν νομίζω ότι είναι υπερβολικό το κανονιστικό πλαίσιο. Νομίζω, όπως σας είπα, πως ήταν αρκετά γενναιόδορη η φάση εφαρμογής διαφόρων μέτρων ακριβώς για να συνεχιστεί η δυνατότητα δανειοδότησης πραγματικής οικονομίας παρά τους πιο αυστηρούς κανόνες. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε, ούτω ώστε οι τράπεζες να αντιμετωπίσουν τις μη εξυπηρετούμενες εκθέσεις για να μπορούν να κάνουν περισσότερες δανειοδοτήσεις στην πραγματική οικονομία. Υπάρχουν διαφορές στο πώς χορηγούνται τα δάνεια στις μικρομεσαίες από χώρα σε χώρα. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Εξαρτάται από την οικονομική κατάσταση της χώρας, τους ρυθμούς ανάπτυξης. Νομίζω ότι η Τραπεζική Ένωση μειώνει αυτές τις διαφορές. Αλλά από μόνη της δεν μπορεί να τις καταργήσει. Αλλά όπως είπατε κι εσείς, κινούμεθα προς την κατεύθυνση της ε, Ένωσης των Κεφαλαιαγορών, το CMU. Αυτό λοιπόν που, που κάνει η, Ευρωπαϊκή, Αγγλική συγγνώμη, Κεντρική Τράπεζα, που προσπαθεί δηλαδή να αναπτύξει πολύ διαφανείς δυνατότητες εξασφάλισης των δανείων, αυτό μπορεί να βοηθήσει και η συλλογή στοιχείων και το Μητρό θα βοηθήσει. Αλλά επαναρχόμαστε στο πρόβλημα που ήδη συζητήσαμε. Μήπως είμαστε υπερβολικοί, μήπως ζητάμε υπερβολικά στοιχεία για αυτό το Μητρό στοιχείων. Θα πρέπει να πετύχουμε τη σωστή ισορροπία. Να δούμε πόσα στοιχεία χρειαζόμαστε από τις τράπεζες, και πόσο μπορούν οι τράπεζες, ιδιαίτερα οι μικρότερες, να μας τα στείλουν. Αλλά αν θέλουμε να χρηματοδοτήσουμε τις μικρομεσαίες, μιλάμε για τις τράπεζες χορήγησης ε, λιανικών υπηρεσιών, που είναι μικρομεσαίες τράπεζες. Και βεβαίως ε, τις επιβαρύνει η αποστολή στοιχείων. Πρόεδρος, ο Νότης Μαριάς. Ευχηθήκατε να υπάρξει λευκός καπνός στις διαπραγματεύσεις της Ελληνική κυβέρνηση με την Τρόικα. Αλλά να σα πληροφορήσω ότι αυτή τη στιγμή η Τρόικα ζητάει και νέα σκληρά μέτρα, ζητάει μειώσει των συντάξεων στην Ελλάδα, ζητάει απολύσει δημοσίων υπαλλήλων και άλλα. Ένα από τα επιχειρήματα που υπάρχουν προ την ελληνική κυβέρνηση είναι ότι αν δεν υπογράψει τη συνέχιση του προγράμματο, τότε δεν θα γίνεται χρηματοδότηση των ελληνικών τραπεζών από τον έκτακτο μηχανισμό, τον ΕΛΑ. Έχω εδώ μία απάντηση που μου δώσατε σε ερώτηση που σας έκανα πριν από αρκετούς μήνες και η απάντηση είναι 2 Απριλίου. Η ερώτηση ήταν για ποιο λόγο είχατε πει στις ελληνικές τράπεζες να μην αγοράζουν T-bills, δηλαδή γραμμάτια του ελληνικού δημοσίου. Από την απάντηση προκύπτει όμως το εξής, ότι λέτε ότι θα υπάρχει ίση μεταχείριση των ελληνικών τραπεζών με τις άλλες τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την εποπτεία. Επομένως η ερώτησή μου είναι απλή. Εάν δεν υπάρξει συμφωνία της Ελλάδας με τους δανειστές της στις 30 Ιουνίου και από την 1η Ιουλίου δεν υπάρχει πρόγραμμα, δεν υπάρχει μνημόνιο, θα υπάρξει καμία διαφοροποίηση από πλευράς Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στη χρηματοδότηση των ελληνικών τραπεζών μέσα από το σύστημα ΕΛΑ. Θα αλλάξουν δηλαδή τα κριτήρια του συστήματος ΕΛΑ παρότι η Ελλάδα δεν θα είναι σε μνημόνιο. Και η εποπτική δράση δικιά σας θα αλλάξει αν η Ελλάδα δεν είναι σε μνημόνιο. Ή μήπως δεν έχει καμιά σημασία για τη ρευστότητα των τραπεζών το ότι η Ελλάδα δεν θα είναι σε μνημόνιο μετά την 30η Ιουνίου. Ευχαριστώ. We collect the last catch the eye question, Και η τελευταία ερώτηση προς προσέχει και κ. Ζαριανόπουλος. Απλώς θυμίζω ότι ήμουνα στον, με απάντηση της γραμματείας σας στον κύκλο των ομιλητών και στη διαδικασία ΚΑΤΣΔΙΑΙ. Τέλος πάντων. Ε, κυρία Πρόεδρε, τη γνώμη σας για τρία θέματα που αφορούν την Ελλάδα, αφού σημειώσω ότι ως επόπτης φερεγγιότητας των τραπεζών συμμετέχετε ενεργά στη διαμόρφωση της πολιτικής για την Ελλάδα, όπως για παράδειγμα την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών στα πλαίσια του μνημονίου που αύξησε το χρέος της χώρας ή τη μετατροπή ιδιωτικού χρέους της χώρας προς ευρωπαϊκές τράπεζες, τη μετατροπή του σε κρατικό χρέος προς κράτη. Στα πλαίσια του μνημονίου ο κόσμος στην Ελλάδα, ο λαός πτώχινε, έμειναν πολύ άνεργοι, δεν μπορούν να πληρώσουν τα δάνεια, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στην Ελλάδα είναι η μεγάλη τους πλειοψηφία. Τώρα έρχονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση και η Τρόικα ζητάει ακόμα περισσότερα, δηλαδή μεγαλύτερη πτώχευση του, του λαού και μεγαλύτερη αδυναμία να ξεπληρωθούν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Ήδη ξεκίνησαν χιλιάδε πληστηριασμοί και ο κόσμο κάνει τα σπίτια του. Πιστεύετε ότι η βιωσιμότητα των τραπεζών την οποία ελέγχεται στην πραγματικότητα εμεί λέμε ότι είναι συμβαδίζει με την πτώχευση, με την εξαθλίωση του κόσμου και ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα όσον αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Δεύτερο ερώτημα. Πολλές ελληνικές τράπεζες έχουν τιτλοποιήσει τα δάνειά τους. Τα πουλάνε σε επενδυτικούς οίκους σε αξία πολύ χαμηλότερη από την πραγματική τους αξία. Οι επενδυτικοί οίκοι με τη σειρά τους ζητάνε ολόκληρη την αξία. Δηλαδή βγάζουν ένα τεράστιο κέρδος με ιδιαίτερα έντονη και ανεξέλεγκτη πίεση για την ίσπραξή τους που έχει οδηγήσει σε πάρα πολλές αυτοκτονίες. Αυτήν τη φερεγγιότητα Και τελευταίο, τη γνώμη σας για την δημιουργία κακής τράπεζας, bad bank, για την ανάληψη των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην ε, Ελλάδα και ποιος θα πληρώσει τελικά τις τράπεζες για να πουλήσουν αυτά τα δάνεια στη λεγόμενη bad bank. Λοιπόν, Καταρχάς να πω ότι έχω κάθε συμπάθεια και κατανόηση για τις δυσχέρειες ε, των Ελλήνων πολιτών σε αυτή τη συγκυρία και να σας πω ότι και σε ιδιωτικές συζητήσεις με τους συναδέλφους μου, τους ε, Έλληνες επόπτες, ε, το συζητάμε λοιπόν αυτό και γνωρίζω λοιπόν πόσο άσχημα είναι τα πράγματα για το λαό. Αλλά εγώ δεν έχω καμία σχέση με τον ELA, τον ειδικό μηχανισμό βοήθειας για την ε, ρευστότητα. Εσείς οι νομοθέτες, εν τη σοφία σας, δημιουργήσατε αυτό το διαχωρισμό μεταξύ νομισματικής πολιτικής και εποπτείας. Και όντως, όταν ε, εξετάζουμε τις ελληνικές τράπεζες, τις αντιμετωπίζουμε, τις αντιμετωπίζουμε όπως ε, οποιαδήποτε άλλη τράπεζα στα πλαίσια του SSM. Ίδια κατάσταση. Τα ίδια κριτήρια εφαρμόζουμε με την μέγιστη ομοιομορφία λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιομορφίες των χωρών και καταστάσεων. Αυτό δεν έχει αλλάξει. Βεβαίως, βεβαίως, εφόσον αποφασίζουμε μέσω του ΣΡΕΠ δηλαδή της ε, διαδικασίας ε, αναθεώρησης και αποτίμησης βλέπουμε πώς γίνεται η προληπτική αποτίμηση. Αλλά αυτό το κάνουν οι Έλληνες συνάδελφοι. Είναι πολύ καλοί επιτηρητές, βλέπουν πώς αναδιοργανώνονται, πώς αναδιαρθρώνονται οι τράπεζες και ο ελληνικός τραπεζικός τομέας. Δεν υπάρχει τίποτα το διαφορετικό εδώ και εργαζόμεθα με βάση τη θαυμάσια εργασία τους, επί της οποίας οικοδομούμε για την ερώτηση για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, έχω πλήρη συνέστηση ότι δεν είναι μόνο τραπεζικό πρόβλημα, ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Όπως είπα και προηγουμένως, θα επιχειρήσουμε να εκτιμήσουμε αν αυτό που έγινε στην Ιρλανδία μπορεί να αξιοποιηθεί, να αξιοποιηθεί ως ε, πρότυπο για άλλες χώρες και για να γίνει αυτό θα ακούσουμε από τους ε, Ιρλανδούς επόπτες που ε, έκανε αυτή τη διαδικασία ναι, να τελειώσω, να τελειώσω η τιτλοποίηση μπορεί να είναι ή όχι μια λύση, εξαρτάται από την περίπτωση. Τώρα για την κακή τράπεζα, ναι, ναι, μπορεί να είναι η λύση μια κακή τράπεζα. Αλλά πρέπει να το δούμε στα πλαίσια του νομικού πλαισίου. Δηλαδή, αν είναι δημόσια κακή τράπεζα, πρέπει να την αποδεχθεί η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Κομισιόν. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Ήταν μια πολύ πλούσια και ενδιαφέρουσα ακρόαση. Η δεύτερη τακτική δημόσια ακρόαση για το 2015 θα γίνει στις 19 Οκτωβρίου. Θα αποφασίσουμε και θα σας ενημερώσουμε έγκαιρα για τα θέματα που θα θέλαμε να δείξετε και τις ερωτήσεις μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Thank you. Sorry, there was a small problem to us. Ευχαριστώ, με συγχωρείτε. Υπήρχε ένα μικρό πρόβλημα με τον κατάλογο ψηφοφοριών. Να προχωρήσουμε όμως αμέσως στην ψηφοφορία. Ξεκινάμε με το κείμενο, με το, το τεστ. Κάρτα ψηφοφορίας. Ε, όποιος δεν έχει, παρακαλώ να σηκώσει το χέρι του. Μόνο η υπερβάνς, μπερές, ωραία, το σημειώνουμε. Ξεκινούμε το τεστ, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Ωραία. Ξεκινούμε με την έκθεση του Sven Giegold για τις στατιστικές για το συγκεκριμένο πληρωμών των Διεθνής εμπόρων Υπηρεσιών και τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Συμβαστική Α σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Έλεγχος για το δεύτερο τμήμα. Άρχεται του ψηφοφορία. Ε. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 22. Υπέρ. Τρεις σελίδες από μετά. Όχι, όχι, καταπίπτουν. 42. Με συγχωρείτε, 22, 22, όπως είπα. 22 υπέρ. Κατά. Ακούγεται να εγκρίνεται. Έλεγχος. Πέρας. 23, 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική B υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική C υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ κατά έλεγχο για τον 27. Άρχεται η ψηφοφορία. Vote is closed. Πέρας. Απορρίπτεται. 28. Δεν θα ψηφιστεί. 4. Υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά ας ελέγξουμε. Περάς. Αγκρίνεται. 29 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 30 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 31 υπέρ, κατά, ελέγχουμε για τα 31, άρχεται η ψηφοφορία. Closed. Yeah, Απορρίπτεται. Μιλάει. 32 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική E υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε για την 8 άρχεται η ψηφορία πέρας εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Ψηφίζουμε το κείμενο όπως τροποποιήθηκε, ονομαστικά, του ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ψηφίζω για το νομοθετικό ψήφισμα. Άρχεται ψηφοφορία, ονομαστικά. Πέρας. Εγκρίθηκε. Απόφαση για δημοκρατική εντολή. Κανονός άρθρος 73. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. ψηφίσει κάποιοι συνάδελφοι. Πέρας. Εγκρίνεται με απόλυτη πλειοψηφία. Σαφή πλειοψηφία μάλλον. Οπότε μπορούμε να περάσουμε σε διαμαρτυρίε με το Συμβούλιο. Ευχαριστούμε και συγχαρητήρια στον εισηγητή. Τώρα περνάμε στο σχέδιο γνωμοδότησης του Γεωργίου Κίρτσου για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία και την χρηστή οικονομική διακυβέρνηση. Συμβιβαστική α υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ κατά επαλήθευση για την 7 άρχεται η ψηφοφορία. έληξε. Εγκρίνεται. Άρα οι 13, 14, 15, 20 καταπίπτουν. 9. Τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά. Ποιες εγκρίνεται. 11. Υπέρ. Κατά. Επαλήθευση για την 11. Άρχεται. Έληξε. Εγκρίνεται. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 13 υπέρ. Α, 15 υπέρ. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 υπέρ κατά νομίζω ότι απορρίφθηκε αλλά θα επαληθεύσουμε τη 18 έληξε απορρίπτεται α, η ισοψηφία Συμβιβαστική Β σε μερικά τμήματα. Λοιπόν, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ Κατά. Επαλήθευση για την 28. Άρχεται. Έληξε. Περέσει υπέρ. Εγκρίνεται λοιπόν. 29 υπέρ. Κατά επαλήθευση και για την 29 άρχεται έληξε πάλι ισοψηφία απορρίπτεται λοιπόν 30 υπέρ κατά δεν βλέπω καλά τα χέρια 30 ξανά α Α, καλά, καλά, εγκρίνεται, εγκρίνεται. Α, ναι, δεν είναι. Συμβιβαστική γάμα, πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική δέλτα, Όχι, πρώτα την 49. Την 39. 39 υπέρ. Κατά. Υπέρ κατά επαλήθευση, επαλήθευση για την 39. 39, 3 και 9. Κολλητά. Έληξε. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική δέλτα με προφορική τροποποίηση. Πρώτα την προφορική τροποποίηση υπέρ. Κατά. Επαλήθευση για την προφορική άρχισε. Έληξε. Απορρίπτεται. Τώρα η συμβιβαστική χωρίς την προφορική τροποποίηση υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 45 υπέρ κατά επαλήθευση Έληξε. Εγκρίνεται. Άρα καταπίπτει 46, 48 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 47 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Το αρχικό κείμενο υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 49 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 53 υπέρ κατά επαλήθευση για την 53 Εγκρίνεται. Συμβιβαστική F με προφορική τροποποίηση. Πρώτα την προφορική υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Εξήντα υπέρ. Κατά αποχές επαλήθευση άρχεται. Έληξε. Εγκρίνεται. Το κείμενο όπως τροποποιήθηκε. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Uh, the vote is concluded and uh... Έληξε η ψηφοφορία. Όπως ξέρετε, λόγω των εξαιρετικών συνθήκων ε, στο Eurogroup, το επόμενο σημείο θα αναβληθεί. Άρα λίγη εδώ η συνεδρίαση η επόμενη την Τετάρτη στις 15 Ιουλίου στις 3 το απόγευμα και την επόμενη μέρα. Ευχαριστούμε λίγη συνεδρίαση.